Ähm, so, ich bin unterrichtet worden, dass wir jetzt den ersten Punkt nicht ohne die Kommission verhandeln. Λοιπόν, μου είπαν ότι δεν μπορούμε να εξετάσουμε το πρώτο θέμα χωρίς την Επιτροπή, που νομίζω όμως ότι εντωμεταξύ ήρθε και μπορεί να τοποθετηθεί, αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να λάβει το λόγο η συγγήτρια. Για το πρώτο ε, σημείο της ε, ψηφοφορία μου είπαν ότι επιθυμεί το λόγο η Γενική Συγήτρια. Oui. Oui. Mais il n'y a pas de rapport à voter, non Ah, ah voilà. Donc, il faut donner la parole à monsieur. Ο κύριος Αντεπρέ είναι αυτός πρέπει να μιλήσει, όχι εγώ. Α, τότε δεν ενημερώθηκα καλά. Ο κύριος Ντεπρέ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε μια μεταφορά κονδυλίων όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής και Παγκοσμιοποίηση. Για τρεις λόγους γίνεται το αίτημα αυτό. Πρώτον, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε τη μεταφορά αυτή προτού εγκρίνουμε την ίδια την έκθεση που αδειοδοτεί, την απόφαση δηλαδή που αδειοδοτεί τη μεταφορά αυτή θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή πριν από τη μεταφορά, καθότι 28 Μαΐου είναι η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς μπορούμε εμείς να ψηφίσουμε τη μεταφορά αυτή σήμερα. Πρώτος στόχος για τον οποίο δεν θέλω να γίνει αυτή τη στιγμή ψηφοφορία. Θα ήθελα να γνωρίζω επίσης προτού προτείνω την δική μου την πρόταση, να γνωρίζω ποια είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την δική της αξιολόγηση για τα τελευταία έτη, δηλαδή ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την χρησιμοποίηση του Ταμείου αυτού τα τελευταία έτη. Κύριε Πρόεδρε, παραλαμβάνω. Αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτού ολοκληρώσω την έκθεση αυτή για την τεχνική υποστήριξη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, θα ήθελα και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι η εξολόγηση που έχει κάνει όσον αφορά τι επιδόσει του Ταμείου αυτού προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση για την παρελθούσα χρονική περίοδο. Χρειάζομαι το έγγραφο αυτό. Και τρίτον, Μία ερώτηση που θέλω να υποβάλω γιατί μου έκανε κάπως εντύπωση μόλον ότι αυτό είναι ίσονος σημασίας μου κάνει εντύπωση στα πλαίσια της μεταφοράς αυτής το ότι ζητάμε αυτή τη στιγμή ήδη για το προπολογισμό του 2015 πιστώσεις για κάποιες συνεδριάσεις οι οποίες είναι καθαρά τεχνικής φύσης και οι οποίες νομίζω ότι δεν δικαιολογούνται και αναφέρονται βασικά στο έτος 2016. Λοιπόν, συνοψίζω πρώτον. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε αυτή τη στιγμή την ελόγω μεταφορά προτού εγκρίνουμε την απόφαση που ιδιοδοτεί τη μεταφορά αυτή. Δεύτερον, θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η εξολόγηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο αυτό προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μου τη δώσει. Και τρίτον, ερώτημα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ε, χρησιμοποίηση πιστώσεων 2015 για τεχνικέ συνεδριάσει που θα λάβουν χώρα μόνο το 2016 και δεν νομίζω ότι ε, θα υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή να εγκρίνουμε αργότερα τη μεταφορά αυτή. Πέρυσι η σχετική μεταφορά είχε γίνει τον Δεκέμβριο. Θα μπορούσαμε εμείς να ψηφίσουμε τον Ιούνιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ähm, λοιπόν, οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις αφορούν την ε, Επιτροπή, την Κομισιόν. Δεν ξέρω αν είναι σε θέση να αντιδράσει. Sorry, I apologize for the delay. We thought that you were having the restricted meeting. Uh. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Νόμιζα ότι είχατε την ε, συνεδρίαση κλεισμένων των θυρών και περίμενα απ' έξω. Ε, il a demandé. Et concernant... Κύριε Ντεπρέ, προφανώς μπορούμε να σας δώσουμε την έκθεση αυτή αξιολόγησης. Εμείς για τις τεχνικές αυτές συνεδριάσεις θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να γίνουν κάποιες προκειμένου να κινητοποιηθεί το ταμείο αυτό. Ενδεχομένως ο συναδελφός μου να μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντω, για να προετοιμαστούν οι συνεδριάσεις αυτές θα υπάρχουν ε, εμπειρογνώμονε και εκπρόσωποι από διάφορε ε, χώρε και θελήσαμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάποιες τεχνικές συνεδριάσεις προκειμένου να δοθούν συγκεκριμένε εντολές και συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής όσον αφορά κάποια προγράμματα. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ήδη από τώρα θα έπρεπε να γίνει ένας προγραμματισμός για το 2016 και προφανώς η μεταφορά αυτή θα μπορούσε να γίνει και κάποια στιγμή αργότερα. Ενδεχομένως να γίνει μεταφορά των κονδυλίων αυτών όταν κινητοποιηθεί και το ίδιο το Ταμείο. Ο κύριος Δεπρέ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να μας απασχολήσουν στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας και σας υπόσχομαι θα κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Έχει Επιτροπή να παρατηρήσει κάτι. Από ό,τι φαίνεται όχι. Άρα δηλαδή <laughs> τώρα έχουμε ένα άλλο πρόβλημα ότι πρέπει να περιμένουμε την κυρία Χόλμαια που μου είπαν ότι έρχεται, αλλά σχετικό είναι και αυτό. Gut, da wir nicht genau wissen... Λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα έρθει η κυρία Χολμάια, ε, προτείνουμε οι δύο ε, ψηφορίες ε, για τις ε, μεταφορές και για την πολιτική των κτηρίων να αναβληθούν. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 6. Στο σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού αριθμός 3 και η γενική συγγήτρια η κυρία Γκατζία Ζαμπάλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να σπω. πω για τον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμού 3 και ακόμα και για τον 4 που από κοινού μπορούμε να το δούμε γιατί η παρουσίαση παρότι δεν έχουν καμιά σχέση το ένα με το άλλο η παρουσίαση έγινε από κοινού του 3 και του 4 των διορθωτικών προϋπολογισμών. Έχουμε προθεσμία κατάθεση τροπολογισμών, ε, τροπολογιών μέχρι τις 5 Ιουνίου η ιδέα είναι να ψηφιστεί στις 23 Ιουνίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να εγκριθεί στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου την περίοδο συνόδου του Ιουλίου. Και αν δεν κάνω λάθος, το ίδιο χρονοδιάγραμμα υπάρχει για τον διορθωτικό προϋπολογισμό 4 ώστε τον Ιούλιο να μπορούμε αυτούς τους δύο διορθωτικούς να τους έχουμε εγκρίνει στην Ολομέλεια. Φαίνεται ότι το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εργάστηκε γοργά και αποτελεσματικά και ενέκριναν τις προτάσεις, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς τροποποίησης Και γι' αυτό <clears throat> αν δεν υπάρξει κάποια οποιαδήποτε περιπλοκή μπορούμε να εγκρίνουμε γοργά αυτούς τους δύο διορθωτικούς προϋπολογισμούς και εμείς. Ο τρία έχει σχέση με το πλεόνασμα το περσινό, το, ο διορθωτικός 4 αφορά το θέμα της αλληλεγγύης όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης και ε, από πλευράς μας αυτό πρέπει να γίνει. Μπορούμε γοργά να προχωρήσουμε νομίζω χωρίς ε, οποιασδήποτε ε, φιλοσοφικές ας το πω έτσι παρεκκλήσεις προς το Συμβούλιο. Παρατηρήσει από αυτού παρακαλώ, από ό,τι βλέπω όχι. Ήρθε η κυρία Χολμάια. Κυρία Χόλμα, μόλις ε, ε, ξεκουραστείτε, πάρτε μια ανάσα μάλλον, ε, μπορείτε να μας ενημερώσετε για τα σημεία 13 και 14. Ωραία λοιπόν. Καταρχήν θα αναφερθώ στις μεταφορές. Η μία είναι μεταφορά του ελεγκτικού συναντρίου, το οποίο κατέρευσε το μηχανογραφικό σύστημα και έπρεπε να ε, επιδιορθωθεί το σύστημα ε, εκβάθρων. 685.000 χρειάστηκαν. Και ελπίζουμε αυτό να μην ξαναγίνει στο ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί τώρα πλέον η υποδομή ε, θα πρέπει να είναι σύγχρονη. Εκεί υπάρχουν και πάρα πολλά ευαίσθητα στοιχεία και για την ασφάλεια αυτών των στοιχείων αρμόδιοι είμαστε εμείς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν εμείς μόνοι μας ε, θεσπίζουμε τόσο πολλούς κανονισμούς για την ασφάλεια των στοιχείων, ε, θα πρέπει τουλάχιστον να φροντίζουμε τα του οίκου μας. Έτσι λοιπόν ε, αυτές τις 685.000 που τις πήραμε από ένα άλλο κεφάλαιο από τους συμβασιούχους ε, θα τις ε, μεταφέρουμε στο κεφάλαιο υπαρθμών 21 εκεί που γίνεται λόγος ε, για τη συντήρηση εξοπλισμών, όπως σας είπα 685.000 είναι το ποσό. Το δεύτερο αφορά στην Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία στο μέλλον θα χρησιμοποιεί τα δικά μας τα κτίρια. Και γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή των Περιφερειών έπρεπε και αυτή να πληρώσει το δικό της το ποσοστό ε, για το προσωπικό ασφαλείας. Αυτό θα το κάνει η Επιτροπή των Περιφερειών και να το κάνει αυτό χρειάζεται επιπρόσθετα 38.000 ευρώ. Και η τρίτη μεταφορά αφορά επίσης ε, την Επιτροπή των Περιφερειών. Κάτι παρεμφερές είχαμε την τελευταία φορά στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Πρόκειται για 15.000 επιπρόσθετα κονδύλια που είναι το αυξημένο κόστος ε, για τον βρεφονιπιακό σταθμό. Αυξήθηκε το κόστος σε 660.000. Μέχρι τώρα υπάρχουν 450.000, γι' αυτό πρέπει να μεταφερθούν 215.000 έτσι ώστε να μπορούμε να καλύψουμε το κόστος που καλύπτει και που καταβάλει το ποσό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ σας καλώ να ψηφίσετε και τις τρεις αυτές μεταφορές. Πρόεδρος, δεν ξέρω, ε, μήπως έχει κάποιος ε, διαφωνία, διαφωνεί κανείς να ε, ψηφίσουμε unblock. Από ό,τι βλέπω όλοι συμφωνείτε να ψηφίσουμε και για τα τρία αυτά θέματα και για τις τρεις μεταφορές και μου είπαν ότι η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά. Παρακαλώ λοιπόν ε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά όποιοι συμφωνεί με αυτές τις μεταφορές κονδυλίων. Okay. Okay. Ja, dann zählen wir die Isabel so mit. Ah, Da ist sie. Okay. Gut. Haben alle abgestimmt.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 θα πρέπει να σας ενημερώσω για το ότι ε, πολύ συχνά έχουμε το πρόβλημα των δύο εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Βρυξέλλες και Στρασβούργο. Και η Ιουλίσα, ο οργανισμός αυτός, έχει και αυτός δύο έδρες, μία έδρα στο Στρασβούργο και μία στο Ταλίνα. Και να συνημερώσω λίγο και για το κόστος. Όταν αγοράζω Στρασβούργο ένα πακέτο Μάλμπορο, και αυτή τη στιγμή δεν κάνω προπαγάνδα για το κάπνισμα, Είναι 7 ευρώ. Στο Ταλίν το αγοράζω για 3 ευρώ και 50 λεπτά. Ενδεχομένως λοιπόν θα πρέπει, δεν θα πρέπει το κτίριο να κτιστεί στο Στρασβούργο, αν μπορεί να ανεργεθεί σε μια άλλη πόλη στο Ταλίν, στο ίμις της τιμής συγκεκριμένα. Συνεπώς συνειδητοποιώ το πρόβλημα που υπάρχει με τις συνθήκες εργασίας στο Στρασβούργο πολλές φορές, αλλά από την άλλη είμαστε προσεκτικοί με το τι αποφάσεις λαμβάνουμε κάθε φορά που φασίζουμε για την έδρα μιας υπηρεσίας ενός εξωτερικού φορέα. Αυτή τη στιγμή δεν επικρίνω κανέναν και ούτε λέω ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να διαχωριστεί ανάμεσα στις δύο τις έδρες ο οργανισμός αυτός. Ευχαριστώ. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει μια μεγάλη συζήτηση, αλλά κυρία Χόλμα έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται συζήτηση γιατί συμφωνώ με τον συνάδελφο και πρέπει να σας πω ότι τα κράτη-μέλη είναι εκείνα τα οποία είναι αρμόδια για την, τον ορισμό των εντρών των περιφερειακών γραφείων. Δεν, μας, ε, συμφώνησαν μαζί μας και εμείς υποχωρήσαμε. Είχαμε πει στην Εστονία, επειδή όμως η αρχική έντρα ήταν στη Γαλλία και οι Γάλλοι ε, διαφώνησαν να συγκεντρωθούν οι, τα γραφεία αυτά στην Εστονία. Εμείς πιστεύαμε Εστονία ε, θα ήταν ε, θαυμάσια έντρα για να πάρει και αυτή έναν οργανισμό ε, το Ιουλίζα. Όλα τα άλλα κτίρια ήταν ήδη στο Στρασβούργο. Τελικά αποφασίσαμε για δύο έδρες και πιστεύουμε ότι επειδή ε, υπάρχει το μηχανολογικό, δεν θα προκύψουν ε, σημαντικές δαπάνες. Ο συνάλφος τώρα πρέπει να ξέρει ότι συμφωνούμε εμείς ως Κοινοβούλιο μαζί του, αλλά δυστυχώς οι έδρες των περιφερειακών οργανισμών ε, έχουν ήδη προκαθοριστεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι διαφωνούμε κάθετα. Ε, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ε, γι' αυτό λοιπόν το θέμα της έντρας σας λέω έχει κριθεί και δεν μπορούμε εμείς τίποτα να κάνουμε επ' αυτού. So, ähm, wir haben jetzt eine... Λοιπόν, διαδικαστικό τώρα. Η κυρία Χολμα, εγώ προτείνω να γνωμοδοτήσουμε όπου θα συμπεριλάβουμε και τη γνώμη του συναντέλφου και μέχρι τις 8 ε, Ιουνίου να αποφασίσουμε οριστικά. Και Ευχαριστώ ε, να στείλω τη γνωμοδότηση και στον Σνάλφο Τάραντα και στον κύριο Ντεπρέ ε, όταν θα έχουμε και τα τελικά στοιχεία. Πρόεδρος, δεν έχω καμία διαφωνία, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντεπρέ. Πρέπει όμως να ξέρετε, από ό,τι με ενημέρωσαν, ότι έχουμε ήδη ε, δώσει μία παράταση. Μισό λεπτό. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Λοιπόν, η γραμματεία με ενημέρωσε ότι αν τελικά δεν υπάρχει διαφωνία στην Επιτροπή και η Επιτροπή Κομισιών ε, δεν διαφωνήσει, μπορούμε να αποφασίσουμε στις 8. Αν όμως θέλουμε να τηρήσουμε αυστηρά τους κανονισμούς, ήδη εξαντλήσαμε τη δυνατότητά μας για παράτηση και πρέπει σήμερα να αποφασίσουμε καταρχήν ο κ. Ντεπρέ και μετά η συγγήτρια. Oui. Euh, Κύριε Πρόεδρε, Ας δούμε λίγο τα πράγματα σοβαρά σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριο Στάραν και θέτω το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά ένα άλλο σύστημα μεγάλης κλίμακας, το SES, e πάλι εκεί πέρα έχουμε δύο έδρες για λόγους ασφάλειας. Από τη μία πλευρά έχουμε έναν εξοπλισμό ο οποίος βρίσκεται στο Στρασβούργο και από την άλλη έχουμε κάποιους άλλους εξοπλισμούς μεγάλης κλίμακας που νομίζω ότι βρίσκεται κάπου στην Αυστρία αν δεν κάνω λάθος. Η ίδια λογική διέπει και αυτόν τον οργανισμό γιατί δεν είναι τόσο χαζός ακούγεται αυτή τη στιγμή. Επομένω, θα ήθελα να γνωρίζω, να μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν η ίδια λογική διέπει και την πρόταση που έχουμε εδώ πέρα για τον ίδιο e Λίζα. Διαφωνώ όμω με αυτά που είπε ο κύριο ε, Τάραν, γιατί να ακολουθήσουμε τη δική του τη λογιστική. Όλα θα πρέπει να πάνε στη Ρήγα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα πρέπει να μα πληρώνουν με το μέσο μισθό τη περιοχή εκείνη. Und Τώρα, από ό,τι φαίνεται, γίνεται πάλι σύντηση που φοβόμουν. Η κυρία Χόλμαρ, αυτά τα οποία έθιξε ο συνάδελφος κ. Τεπρέ αφορά τον σερβερ στην Αυστρία, ε, που δεν μπορεί όμως να είναι στον ίδιο χώρο, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, αν έχετε ένα τέτοιο σερβερ που είναι για λόγους ασφαλείας, ε, πρέπει να είναι σε κάποιο άλλο χώρο. Αυτό τέλος πάντων δεν είναι στο Στρασβούργο, είναι στην Αυστρία και για το λόγο αυτό υπάρχει αυτή η δεύτερη έδρα. Στη Γαλλία και την Εστονία, η Γαλλία δεν ήθελε να παραιτηθεί του Στρασβούργου, η Εστονία έπρεπε να πάρει αυτόν τον οργανισμό και γι' αυτό το λόγο ε, σας λέω προέκυψε αυτή ο μισοσυμβιβασμός. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε δυστυχώς ε, αυτό το συμβιβασμό και όσον αφορά τον κανονισμό θέλω να πω ότι αν αποφασίσουμε σήμερα να ε, γνωμοδοτήσουμε τότε μπορούμε να ψηφίσουμε μετά από δύο εβδομάδες. Πρόεδρος, δεν θα ξεκινήσουμε τώρα επίσημη συζήτηση. Ολόκληρη συζήτηση, γιατί νομίζω θα μας χαλάσει το απόγευμα. Και ε, ρωτώ, ε, υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με την ε, πρόταση της κυρίας Χούλμα να αποφασίσουμε στις 8 εκτό, όχι. Υπάρχει ε, διαφωνία από πλευράς της Κομισιόν επί του θέματος. Αυτό το αποφασίζει η Κομισιόν, όχι ο κύριος Ντεπρέ. Kommission berät Πρόεδρε, θέλω να πω να υπάρχει περιορισμός στο χρόνο όσον αφορά τις υποχρεώσεις της Επιτροπής ε, και του οργανισμού εμείς ε, με μεγάλη, μεγάλη μας χαρά να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις Άρα μην ξεχνάτε και τα πρακτικά στοιχεία που έχουν σχέση με την καθυστέρηση. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τοποθετηθεί θετικά ε, και μετά ίσως οι αρμόδιοι μπορούν να τοποθετηθούν και γραπτά. Αυτή είναι ίσως μια κάποια λύση. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, λέει ο Πρόεδρος. Η συγγήτρια παρακαλώ επ' αυτού. Κοιτάξτε, θα έπρεπε να πω ναι, πριν οι συνάδελφοι όμως γνωρίζουν το περιεχόμενο. Και οι σκιώδεις συγγητές νομίζω δεν συμφωνούν απόλυτα με αυτό. Ίσως ε, να πω ότι κοιτάξτε, σε επίπεδο αρχής ε, νομίζω είμαστε όλοι ε, θετικοί. Δηλαδή δεν έχουμε πρόθεση να μπλοκάρουμε όλο αυτό το project, αλλά υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε σχέση με το ε, κόστος το που θα κοστίσει αρχιτεκτονικά. Ε, αυτό δεν απαντήθηκε. Θα ήθελα έτσι να γνωρίζω λιγάκι το κόστος από αρχιτεκτονική σκοπιά για να γνωρίζουμε κατά πόσον έχει γίνει καλός προγραμματισμός αυτού του έργου. Πρόεδρος, κατόπιν τούτου προτείνω το εξής η συγγήτρια έχει δίκιο και ε, συμφωνούν και οι σκιώδεις. Νομίζω λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο όταν ζητάει πληροφορίες να τις παίρνει τις πληροφορίες και μετά να αποφασίζει. Εγώ λοιπόν προτείνω να μετατεθεί η ψηφοφορία για τις 8 έκτου. Συμφωνεί η Επιτροπή. Από ό,τι βλέπω συμφωνείτε όλοι, άρα εγκρίθηκε αυτή η πρόταση. Ε, και έτσι λοιπόν ε, πλέον ολοκληρώσαμε με τις ψηφοφορίες και χρειαστήκαμε και λιγότερο χρόνο από ό,τι είχε αρχικά προβληθεί. Mes chers collègues, συνάδελφοι, σα ζητώ συγγνώμη, διότι έπρεπε να παραστώ σε μια συνεδρίαση στην οποία ήταν παρόν ο ίδιο ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είχε σχέση με του βασικού προσανατολισμούς και τα βασικά συμπεράσματα όσον αφορά τον τριμερή διάλογο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και έφτασα με καθυστέρηση. Κύριε Γκάιερ, σας ευχαριστώ πολύ που με αντικαταστήσατε. Όσον αφορά τώρα την ψηφοφορία, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία και συνεπώς περνάμε στο 14, όχι το καλύψαμε και αυτό, πολύ ωραία. Καλύψτε επίσης το διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 3 και των υπαριθμών 4, πολύ ωραία, την κινητοποίηση του Ταμείου. Άρα είστε στο σημείο 9, σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού αριθμός 5, η κυρία Γκαρτία Μπάλ Ζαμπάλη το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, προτιμώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει πρώτη αυτό το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού. Πολύ ωραία, το λόγο λοιπόν είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Καλβίνιο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι σήμερα έχουμε αρκετά σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών και καλωσορίζω την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτόν που αφορά την Ευρωπαϊκή Μερίσια διάταξη θεματολόγια για τη μετανάστευση. Κατά Μάιο ενέκρινε ένα διορθωτικό προϋπολογισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προτείνει σημαντική ενίσχυση αρκετών κονδυλίων για την υποστήριξη των δράσεων που εκτίθενται στην δήλωση που αφορούσε το έκτακτο συνέδριο ε, του Συμβουλίου κατά την 23η Απριλίου και το ψήφισμα της 29ης Απριλίου του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή ενίσχυση μιας κοινή δράσης Τρίτονα και Ποσειδώνα με την συμμετοχή ε, και των ε, δράσεων άλλων κρατών μελών που χρηματοδοτείται και συντονίζεται από την Frontex. Δεύτερον, να αυξηθεί η έκτακτη βοήθεια που δίνεται σε σχέση με την, ε, τα κονδύλια, με τις δράσεις όπως εντοπισμό, ταυτοποίηση, παροχή ιατρικής βοήθειας και την, ε, ένα σύστημα ανακύκλωσης και επιμερισμού ε, προσφύγων για την εγκατάστασή τους. Ένα σύστημα για την ε, άμεση γοργή επιστροφή μεταναστών και την αντιμετώπιση θεμάτων σε σχέση με το κέρας της Αφρικής και το, τη Βόρεια Αφρική. Το συνολικό ποσό θα είναι 89 εκατομμύρια ανάληψης υποχρεώσεων Ωστόσο όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να κάνουμε χρήση εκείνων που μπόρεσαν να ανακτηθούν ε, σε σχέση με το παρελθόν όσον αφορά προγράμματα για τη διαχείριση συνόρων κτλ. Για αυτούς τους λόγους ε, υπό το διορθωτικό προϋπονισμό 5, 75,8 θα είναι τα εκατομμύρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Το 2015 είναι 76,6 εκατομμύρια. Εξίσου εντοπίσαμε διαθέσιμα κονδύλια και ε, νέα χρήση, πράγμα το οποίο μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τα, τις ανάγκες και Ταυτόχρονα οι πιστώσεις υποχρεώσεων σε σχέση με το πρόγραμμα Γαλιλαίου δεν θα ε, χρησιμοποιηθούν πλήρω. λόγω του ότι υπήρξε καθυστέρηση όσον αφορά την προμήθεια δορυφόρων μέσω τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Και έτσι τώρα για το 2016 αναβάλλονται αυτέ οι δράσει. Θα υπάρχουν λοιπόν αρκετά κονδύλια για την αντιμετώπιση των αναγκών μετανάστευση χωρίς να έχουμε χρήση του περιθωρίου πληρωμών. Αυτό θα έχει λοιπόν, ε, ε, α το θα είναι ουδέτερο από πλευράς ε, δημοσιονομικής. Επίσης η ενίσχυση των στελεχών στις υπηρεσίες, λυπούμε για το ότι αποχώρησε η κυρία Χολμάγερ βέβαια και αύξηση σε σχέση με τις δράσεις. Ιδιαίτερα 23 προσωρινοί υπάλληλοι για την Frontex οι περισσότεροι από αυτούς αλλά επίσης και για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου, καθώς επίσης και για ε, συναφείς δράσεις. Θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή τη σύντομη παρουσίαση τονίζοντας ε, πόσο πιστεύουμε ότι μια γορχή έγκριση αυτού του προϋπολογισμού, διορθωτικού προϋπολογισμού θα απέστελε ένα σωστό μήνυμα προς τα έξω. Είναι επίγουσα προτεραιότητα το θέμα της μετανάστευσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κατανόησε αυτό το Συμβούλιο και ήταν πολύ θετική η αντίδραση. Θα ήταν λοιπόν ένα πολύ θετικό μήνυμα αν το Κοινοβούλιο εξίσου υποστήριζε αυτό τον διορθωτικό προϋπολογισμό ώστε να μπορέσουμε να διαθέσουμε αυτά τα κονδύλια για τις πιστώσεις υποχρεώσεων για τις ανάγκες αυτές. Ευχαριστώ. Merci, madame. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Γκαρθιά Θαμπάλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση αυτού του διορθωτικού προπολογισμού. Θα ξεκινήσω εκεί που σταμάτησε κυρία Καρδίνιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό βλέπει ότι υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη έγκρισης του διορθωτικού προϋπολογισμού και τουλάχιστον εν μέρη να διατεθούν κονδύλια για την μερική αποσυμφόρηση και ανακούφιση των προβλημάτων στη Μεσόγειο και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ε, γοργά να προχωρήσουμε και να εγκρίνουμε ένα διορθωτικό προϋπολογισμό μέχρι τον Ιούλιο ήδη έλαβε το σχέδιο, η Επιτροπή σχέδιο έκθεσης που παρουσιάστηκε για αυτό τον ε, διορθωτικό προϋπολογισμό που ουσιαστικά έχει δύο άξονες. Πρώτον, αληθεύει ότι δεν θα χρειαστεί αυτά τα κονδύλια πληρωμών ο Γαλιλαίος λόγω των καθυστερήσεων σε σχέση με τους δορυφόρους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά αυτή η δυνατότητα αυτών των κονδυλίων μέσα στο πλαίσιο της χρηστής ε, οικονομικής διαχείρισης, διακυβέρνησης. Και όταν θα χρειαστούν αυτά τα κονδύλια θα διατεθούν όταν θα υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Και δεύτερον, αν αληθεύει σε σχέση με την παρουσίαση του ε, συμπληρωματικού προϋπολογισμού για την υπηρεσία ασύλου, για την Frontex και τα λοιπά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και από πλευρά ε, του Ευρωκοινοβουλίου εργαζόμαστε όχι από πλευρά ε, δημοσιονομική μόνο, αλλά στο πολιτικό πλαίσιο, δίνοντα, ε, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα, για να δούμε αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν επαρκούν ή όχι. Και έχουμε την εντύπωση ότι αυτά τα οποία έχουν εγγραφεί εδώ, ναι μεν βαίνουν καλώ, αλλά μελλοντικά μπορεί να, υπάρξει, να υπάρξουν μεγαλύτερες ανάγκες και να χρειαστούν περισσότερα κονδύλια. Είναι ένα σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο γοργά τώρα τίθεται, παρουσιάζεται και πρέπει με την κατάθεση τροπολογιών προς έγκριση και τα λοιπά να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μέχρι τον Ιούλιο. με τη δυνατότητα αυτή κατάθεσης τροπολογιών θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και αν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ΛΥΜΕ, έχουν κάτι να πούν ή κάτι να σχολιάσουν σε σχέση με αυτά. Αν εγκρίνουμε αυτούς, ε, αυτές τις διορθωτικές προτάσεις, τον 5, τον 4 και τον 3 μέχρι τον Ιούλιο, θα είναι μεγάλη είδηση αυτή. Θα είμαστε, ας το πω έτσι, με καθαρά χέρια θα έχουμε ολοκληρώσει σε σχέση με τις ανάγκες του προϋπολογισμού και θα είναι πολύ ευχάριστη η κατάσταση. Και αν καταλήξουμε σε συμφωνία μπορούμε να εγκρίνουμε και τον διορθωτικό προϋπολογισμό 1 και να φωσιωθούμε στις διαπραγματεύσεις εξετάζοντας τις μελλοντικές πλέον προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση και να πω Καταρχάς ότι συμφωνώ απόλυτα με το ότι θα πρέπει γρήγορα να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα όσον αφορά τόσο τη μετανάστευση όσο και το άσυλο. Να θέσω όμως κάποια ερωτήματα πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτον. Όσον αφορά τη Frontex, 26 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον, εκατομμύρια ευρώ επιπλέον και μας λέτε ότι θα τριπλασιάσετε αυτό το ποσό. Όταν μιλούσαμε για την επιχείρηση τρίτων, είπαμε ότι απορροφούσε το 1 τρίτο της Mare Nostrum. 9 εκατομμύρια ευρώ το μήνα κόστιζε το Mare Nostrum, επομένως δίνετε εσείς μόνο 3 εκατομμύρια μηνιαίως αυτή τη στιγμή με το τρίτον. Αν τριπλασιάσετε, τότε χρειάζεστε 42 ουσιαστικά εκατομμύρια. Ή έχει γίνει κάποιος λάθος στον υπολογισμό. Εγώ σε αυτό το ποσό καταλήγω. Άρα πώς καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τριπλασιάζεται το ποσό της Frontex σε σχέση με τα ποσά που δίνονται και το τρίτον. Γιατί προσθέτουμε τώρα και τα ποσά του Ποσειδών. Ενώ το Mare Nostrum αντιστοιχούσε μόνο σε επιχειρήσεις, ε, της επιχείρησης τρίτων. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν πώς καταλήγουμε σε αυτό τον τριπλασιασμό του αρχικού προπολογισμού, γιατί εγώ καταλήγω σε άλλο ποσό. Δεύτερον, συμφωνώ ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα. Θέτω απλώ κάποια ερωτήματα. Δεν αποδοκιμάζω την πρωτοβουλία σε καμία περίπτωση. Συμφωνώ ότι πολύ γρήγορα θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα τη μετανάστευση και του ασύλου που είναι ζητήματα στρατηγική σημασία. Για να καταφέρουμε να ενισχύσουμε το προσωπικό της Frontex, της Ευρωπόλ και της ΕΑΖΟ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, 24 επιπλέον ανθρώπους πρέπει να προσλάβουμε από ό,τι βλέπω. Και καθότι θα πρέπει να μειώσουμε παράλληλα τον αριθμό του προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τι συμπέρασμα πάλι καταλήγουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνονται υπόψη στου γενικούς υπολογισμούς στα νέα άτομα που θέλετε να προσλάβετε, ή τελικά τα άτομα αυτά θα προσληφθούν, αλλά παράλληλα θα διατηρήσετε τη γενικότερη μείωση που πρέπει να υπάρχει όσον αφορά το ενωσιακό προσωπικό. Φαντάζομαι λοιπόν ότι αν υπάρχουν επιπλέον δαπάνε αυτή τη στιγμή δεν κάνετε απλώ ανακατανομή των διαπανών, από κάπου πρέπει να βρείτε τα χρήματα πώς θα γίνουν συμβατά αυτά τα δύο, μείωση και αύξηση παράλληλου του προσωπικού. Τέσσερι επιπλέον πρόσθετε θέσει προβλέπεται για την ΑΖΟ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη για το Άσυλο. Εγώ είδα τη νομική βάση που επιτρέπει στην ΑΖΟ να εργάζεται και λέτε εδώ τέσσερι πρόσθετε θέσει για την αποδιοργάνωση των δικτύων εμπορία ανθρώπων. Μα η ΑΖΟ δεν κάνει τίποτα για αυτά τα δίκτυα εμπορία ανθρώπων. Δεν είναι δική τη αρμοδιότητα κατά πολέμησή του. Ολοκληρώστε κύριε λέει ο Πρόεδρος. Ναι, τρία ερωτήματα είναι, όχι παρατηρήσεις, ούτε επικρίσει. Τρία ερωτήματα που απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα εγώ νόμιζα ότι το τελευταίο σημείο ήταν απλώ μια διαπίστωση, όχι είναι ερώτηση, λέει ο κύριο Ντεπρέ. Κυρία Χολμάιερ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριο Ντεπρέ. Να πω λοιπόν το εξή ότι σε επίπεδο αρχή συμφωνώ το ότι γίνεται ένα βήμα προς τα εμπρός. Το τελευταίο βήμα θα γίνει στο κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα ΣΥΛΟΥ και θα υπάρξει ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης. Αφενός θα προσφερθεί βοήθεια στις ιδιαίτερα θυγόμενες χώρες και δεύτερον θα υπάρχει ένα σχέδιο επαναγκατάστασης ή επαναπρόθεσης. Αυτό που πρέπει όμως να πω είναι το εξής ότι ένα μεγάλο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον τομέα βοήθεια στη Βόρεια Αφρική με την έννοια το να υπάρχει ένα εύρυθμα ε, λειτουργούν σύστημα χωρίς ασύλου ή προστασία των συνόρων ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν τελείως διαφορετικό αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο δεν θα τρομάξει κανένα. Δηλαδή το να ε, προβλεφθούν άλλοι τέσσερις άνθρωποι για τη Βόρεια Αφρική, αυτό θα μας ε, βοηθήσει στο να κάνουμε ένα άλμα προς τα εμπρός. Ε, ερωτώ, λέει η κυρία Χόλμα ηρωνικά, Κοιτάξτε, οι ίδιε τέσσερι θέσει του χρόνου θα καταργηθούν. Άρα δηλαδή τι εννοείται ότι θα τους χρειαστούμε ε, για μόνο τέσσερις ε, μήνες ε, και του χρόνου θα γίνει ένα πραγματικό βήμα προς τα Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι στην Europol. Προβλέπονται άλλες τρεις νέες θέσεις πριν τρομοκρατηθεί κυριολεκτικά το οργανωμένο έγκλημα. Αυτοί οι τρεις επιπρόσθετοι άνθρωποι θα οδηγήσουν σε μια ουσιαστική βελτίωση του αγώνα κατά του δουλεμπορίου. Και αυτοί θα ασχοληθούν ε, με την Αφρικανική Πύρο και την Ευρώπη. Ε, κοιτάξτε, λυπάμαι που είμαι τόσο κοινική και σαρκαστική. Ξέρω ότι για την Europol ε, θα προσθεθεί ένα μόνο άτομο και διαρωτώ με κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εννοεί σοβαρά όλα αυτά που λέει γιατί ας μην ξεχνάμε, βιώνουμε μία τραγική κατάσταση ή κατά πόσον θέλουμε να προχωρήσουμε με αυτά τα πολύ μικρά βήματα και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο από το ε, να σαρκάζω την κατάσταση. Ε, το, η Europol το μόνο το οποίο έχει κάνει είναι να έχει εξοπλίσει τρία νέα κέντρα. Έχουμε λοιπόν την τεχνολογία, δεν έχουμε όμως προσωπικό ή εμπαστέως δεν ξέρουμε πώς να συνδυάσουμε την τεχνολογία με το προσωπικό. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ. Στους, και αυτή είναι μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Θέλετε πραγματικά να ασχοληθούμε με τους ε, τομείς ε, που έχουν ανάγκη είναι η Άσο, είναι η Frontex και η Europol. Εκεί λοιπόν έχουν γίνει σημαντικές ανακατατάξεις και παράλληλα τίθεται και το ερώτημα κατά πόσο η Κομισιόν είναι πρόθυμη επειδή στο νέο προϋπολογισμό ε, θέλει να έχει και αυτή κάποιες επιπρόσθετες ε, θέσεις για την ίδια, είναι πρόθυμη λοιπόν η Επιτροπή να δεχτεί ανακατατάξεις. Εκεί όπου ε, δεν είναι πολύ μεγάλες ανάγκες, εκεί μπορεί να κάνει λίγο πίσω και να δεχτεί άλλες σημαντικότερες ανακατατάξεις τομείς όπου πραγματικά υπάρχει τεράστια κρίση. Σας ευχαριστούμε κυρία Χολμάιερ. Τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ασχολείται με κάποια ζητήματα, αφήνει όμως ε, κάποια άλλα ζητήματα. Μήπως χάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία μας. Αν είναι να προχωρήσουμε συνήμετρα, τότε καλύτερα να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί α, αν υλοποιήσουμε τελικά η ημίμετρα, δίνουμε βάση με επιχειρήματα σε όλους αυτούς που επικρίνουν τελικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δράση της. Η κυρία Γκρέσλερ έχει το λόγο. Μόνικα, επειδή μιλάμε για το προσωπικό, θέλω να ρωτήσω τη Γενική Διευθύντρια τι ακριβώς θα γίνει με τις θέσεις στη Γενική Γραμματεία. Ακούω ότι οι αντιπρόεδροι θα πάρουν ε, θέσεις και γι' αυτό λοιπόν ερωτώ ε, πότε θα γίνει σχετική ενημέρωση. Και δεν ξέρω, αυτό μπορεί να το κάνει μόνη της η Κομισιόν, αλλά υπάρχει και η προϋπόθεση μείωση προσωπικού κατά 5%. Άρα όταν θέλουμε κάπου να αυξήσουμε το προσωπικό, καλό θα ήταν να μας ενημερώσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, άλλες ερωτήσεις. Εγώ έχω μια ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, ο κύριος Αλή, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Είναι νομίζω σωστή χρονική στιγμή, μια και είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση με την, με την πίεση των μεταναστευτικών κυμάτων, πίεση που ουσιαστικά επικεντρώνεται στα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ερώτηση έχω. Δεν είναι απόλυτα σαφές για μένα πώς ακριβώς οι εξωτερικές εντός εισαγωγικών χώρες θα καθορίζονται εκείνες οι χώρες, εκείνα τα κράτη που βρίσκονται κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα επιμεριστούν τα κονδύλια μεταξύ αυτών των εξωτερικών εντός εισαγωγικών χωρών. Όταν συζητούσαμε τις ροές τις μεταναστευτικές μέσα στο πλαίσιο αυτών των προσεγγίσεων είχαμε και ερωτήματα προς την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και προς τις, τους άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες της Ένωσης για τα κριτήρια με βάση τα οποία θα κατανεμηθούν τα κονδύλια Συμφωνούμε βέβαια ότι αυτή τη στιγμή πράγματι πρέπει να παρασχεθεί υποστήριξη, ότι χρειάζονται πρόσθετα κονδύλια. Εντάξει, όμως χρειάζεται μια συνολική ανάλυση για τον επιμερισμό των κονδυλίων σε σχέση με τα κονδύλια που θα είναι διαθέσιμα στο μέλλον. Ποια είναι τα κράτη-μέλη κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων που θα υποστηριχθούν και με βάση ποια κριτήρια θα τύχουν αυτών των κονδυλίων. Ευχαριστώ. Alors Ενδεχομένω να μα δοθεί μια πολύ ευχάριστη έκπληξη αύριο το πρωί, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μα παρουσιάσει το σχέδιο προπολογισμού για το 2016. Μπορεί να είναι απλώ ευσεβή πόθο. Πάντως, μια ερώτηση έχω και εγώ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προβλέπετε εδώ πέρα νέες θέσεις για τη Frontex με έδρα στη Βαρσοβία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν μια σύμβαση μεταξύ Frontex και Πολωνίας. Μήπως θα έπρεπε να διορθωθεί πρώτα αυτό το ζήτημα, πρώτο κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Κυρία Καλβίνιο, μπορείτε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Σε κάθε περίπτωση Είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε και γραπτώς περισσότερες πληροφορίες για να απαντήσουμε πληρέστερα στις ερωτήσεις εκείνες που ενδεχομένω να μην καταφέρουμε να καλύψουμε σήμερα. Για παράδειγμα, το τελευταίο αυτό ερώτημα του κυρίου Αλή, πώς θα καθορίσουμε ποιε είναι αυτέ οι λεγόμενε εξωτερικέ χώρε και πώ θα χρηματοδοτηθούν. Δεν έχω λεπτομερεί πληροφορίε προ αυτό. Θα συνομιλήσω πάντω με του συναδέλφου μου και θα σα δώσουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Ξεκινώντα με την ερώτηση του κυρίου Ντεπχέ προτείναμε να ενισχύσουμε την προπολογισμό, τον προπολογισμό του Frontex με περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ, τόσο σε υποχρεώσει όσο και σε πληρωμές, και αυτό για να καταφέρουμε να ελοποιήσουμε τις κοινέ επιχειρήσεις Τρίτων και Ποσειδών τους τελευταίους μήνες του 2015. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καλύψουμε στα πλαίσια της επιτήρησης το πεδίο που κάλυπτε στο παρελθόν η επιχείρηση Mare Nostrum. Βέβαια το 2015 και το 2016 θα πρέπει να ληφθούν από κοινού υπόψη προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτό τον τριπλασιασμό που προβλέπεται. Ένα μέρος της ενίσχυσης της χρηματοδοτικής θα δοθεί το 2015 και ένα συμπληρωματικό μέρος της ενίσχυσης θα δοθεί το, 2016. Όσον αφορά την ΕΑΣΟ, διάβαζα λίγο ποιε είναι οι αρμοδιότητε τη υπηρεσία αυτή και εγώ θεωρώ ότι πραγματικά έχει μια σχετική αρμοδιότητα και ότι όντω μπορεί μέσω τη επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων να βάλει κατά των δικτύων εμπορία των ανθρώπων. Πάντω μπορώ να σα δώσω πάλι περισσότερε πληροφορίε για το πώ ο οργανισμό αυτό ανταποκρίνεται στου στόχου μα. Να απευθυνθώ τώρα στην κυρία Χολμάιερ και στην κυρία Γκρέσλερ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια κάποια αγανάκτηση και μια κάποια ηρωνία στα σχόλια της κυρίας Χολμάιερ όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή των προτάσεών μας και όσον αφορά το ότι είναι δυσανάλογο τελικά με τους στόχους και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ξεκινάμε όμως με έναν κοινοτικό ενωσιακό προπολογισμό, ο οποίο είναι σχετικά περιορισμένο και καλούμεθα από την άλλη να είμαστε αρκετά φιλόδοξοι. Επομένω, προσπαθούμε να δούμε μέχρι τα τέλη του 2015 και το 2016 τι μπορούμε να πετύχουμε και δυνατόν όσο να τον πιο γρήγορα ιδίω στα πλαίσια του περιορισμού που προβλέπει το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Για το 2015 προβλέπουμε κάποια μέτρα τα οποία θα αντικατοπτρίζονται και στο σχέδιο προπολογισμού του 2016 και ελπίζουμε ότι όντως αύριο θα έχετε ευχάριστα χαρμόσυνα νέα, κύριε Πρόεδρε, και δεν θα είναι βέβαια πλέον έκπληξη γιατί στο αποκάλυψα τώρα. Αλλά θα δείτε συγκεκριμένα στον προπολογισμό αυτό ποιε είναι και οι πολιτικέ μα προτεραιότητε και πώ χρηματοδοτούνται. Όσον αφορά τις θέσεις που προτείνουμε για τις ε, υπηρεσίες αυτές, στόχος μας είναι να βρίσκονται εκτός του γενικότερου στόχου του 5%, της μείωσης 5% στο προπροσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό διότι θεωρούνται σημαντικές οι θέσεις αυτές και θεωρούμε ότι γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να προσμετρηθούν στη γενικότερη μείωση του προσωπικού. Ορισμένα από τα αυτά έρχονται από τις ίδιες τις υπηρεσίες και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη μετανάστευση. Μία από τις υπηρεσίε αυτές ζήτησε επιπλέον προσωπικό για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της ρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο. Αυτό δεν σχετίζεται άμεσα βέβαια με το ζήτημα το οποίο συζητάμε σήμερα, μετανάστευση και άσυλο. Όσον αφορά την εσωτερική τώρα οργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ξέρετε η Επίτροπος Γεωργίεβα κάνει μια γενικότερη αναθεώρηση προκειμένου να πετύχουμε εξοικονόμηση πόρων και καλύτερη κατανομή των πόρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέποντας μείωση δαπανών στους τομείς εκείνους που είχαν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και που ενδεχομένω δεν αποκρίνονται πλέον στι προτεραιότητε που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα από του τομεί ο οποίο θα υποφεληθεί από την ακατανομία αυτών πόρων τι επόμενε εβδομάδε και του επόμενου μήνε είναι ακριβώ ο τομέα αυτό που σχεδίζεται άμεσα με τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευση. Οι σχετικέ δηλαδή γενικέ διευθύνσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να ενισχυθούν σημαντικά τους επόμενους μήνες του 2015. Θα σας δώσουμε λοιπόν περισσότερε πληροφορίες για τις τρεις αυτές υπηρεσίε, για τα τρία αυτά σημεία τα οποία τόνισα, τριπλασιασμός του προπολογισμού για τον τρίτον και τον πρόγραμμα Ποσειδών, περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την κατανομή των πόρων και περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις αρμοδιότητες της ΕΑΖΟ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και σα ζητώ συγγνώμη, αλλά όσον αφορά την κατανομή αυτή σχετικά με την ε, Γενική Γραμματεία, δεν μου απαντήσατε. Το μόνο που μου είπατε είναι ότι η κυρία Γεωργίευα κάνει μία ανάλυση. Πότε προβλέπετε να δημοσιοποιηθεί η ανάλυση αυτή και πότε θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Καλβίνιο, μάλλον η κυρία Χολμάιερ πρώτα έχει κάποια ερώτηση. Έχω κάτι να ρωτήσω. Όταν λέτε ότι υπάρχουν τέσσερι τρεις θέσεις για τη Europol και οι τέσσερις για την ΕΑΖΟ και θα βγουν από το pool της redeployment ανακατάταξη. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι οι τρεις ε, εξαιρούνται από τις περικοπές του 5% ή οι τρεις, οι Frontex και οι άλλοι δύο εξαιρούνται από αυτό το πουλ. Γιατί αυτό θα ήταν ένα τρίκ, δηλαδή να μας λέτε δίθεν ότι εξαιρούνται αυτοί οι οργανισμοί, ε, κατ' ουσίαν όμως ε, εξαιρούνται μόνο αυτές οι θέσεις ε, που σημαίνει 0,01 προσωπικό. Έτσι και αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο ε, παρά να πούμε στις, ε, ε, στους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν αυτοί μόνοι τους τα θέματα του προσωπικού. Εν πάση αυτό δεν θα επηρεάσει καθόλου τα θέματα των απολαβών. Κύριο Δεπχέ, αν κατάλαβα καλά την κυρία Καλβίνιο, το προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί για νέες αποστολές, για νέες επιχειρήσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Το προσωπικό αυτό λοιπόν δεν θα επηρεαστεί από, την γενικό, το γενικότερο στόχο μείωσης 5%. Αυτό ισχύει λοιπόν για τη Frontex, για την Ευρωπόλ και για την ΕΑΖΟ. Και θυμάμαι μια συζήτηση που είχαμε κάνει όσον αφορά το προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όσον αφορά το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν εμεί παίρνουμε επιπλέον προσωπικό για την ασφάλεια και για το cyber security, αυτό φαντάζομαι όμω ότι δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ισχύουν ουσιαστικά διαφορετικοί κανόνε. Κύριε Γκάιερ, θέλετε το λόγο. be on, I wanted to be on the speakers list. Vous voulez intervenir Monsieur okay. Pardon. Also, ο κύριος Γκάια, ε, κοιτάξτε, όλα αυτά τα θέματα που έφτιαξαν η κυρία Χόλμπαν και ο κύριος ε, Ντεπρέ, θέλω να πω τεξί, ότι μπορούμε λιγάκι να το συνεχίσουμε το θέμα, αν θέλετε, αγαπητή Γενική Διευθύντρια. Κατ' ουσίαν όμως πρόκειται για το εξής. Υπάρχει αυτή η ιδέα του redeployment pool <clears throat> όπως την προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή θα πρέπει να κρυθεί αποτυχημένη. Γιατί έχουμε μια κατάσταση όπου για διάφορους λόγους έχουμε νέους περιφερειακούς οργανισμούς που πρέπει να επεκτατούν γιατί αυξάνεται και η σημασία τους. Και αυτό δεν το έχουμε θίξει. Έχουμε δηλαδή οργανισμούς, αυτούς για τους οποίους κουβεντιάζουμε τώρα, ε, των οποίων διευρύνεται το πολιτικό του πεδίο γιατί αυτό το απαιτεί η κρίση. Και Κατά τα άλλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να ακολουθεί μία προσέγγιση που λέει 5% περικοπές, αυτό που συμφωνήθηκε στη Διοργανική Συμφωνία. Αυτό όμως θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση των οργανισμών και νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή, οι εκθέσεις των οργανισμών που μου έχουν υποβληθεί ε, είναι πάρα πολλές ε, και παρουσιάζουν και αυτές αυτό το παράδοξο, αυτά τα πολύ περίεργα που έθιξαν και οι συνάδελφοί μας και εγώ αν θέλετε μπορώ να συνεχίσω την κουβέντα, την βρίσκω πάρα πολύ διαδεσκεδαστική. Όμως τελικά δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε να ασχοληθούμε με αυτό το redeployment, κυρίως σε σχέση με το ELISA, γιατί απλά αυτό το redeployment pool δεν λειτουργεί. Και ο μόνος οργανισμός από τους τρεις που θέλει οπωσδήποτε να τηρήσει αυτό το σχέδιο είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς ως Κοινοβούλιο δεν το θέλουμε. Το Συμβούλιο ε, είπε ότι το 5% όπως το παρουσιάζει η Κομισιόν είναι το ίδιο, μόνο που αυτοί το προτιμούν, το προτιμούν οπωσδήποτε και δυστυχώς τους ε, ε, απατάει πραγματικότητα. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, να πω στον εισηγητή ότι καλύτερα να δούμε λιγάκι το παράδειγμα, να δούμε αυτά τα οποία έχουμε εξετάσει και θέλουμε να εξετάσουμε σχετικά με τον προπολογισμό των οργανισμών για το 2016, να συζητήσουμε μαζί τους και κάπως να βρούμε πάνω σε αυτό μια λύση. Πολύ ωραία. Κυρία Καλβίνιο, μπορείτε να μας διαφωτίσετε περιληπτικά για όλα αυτά τα ζητήματα. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε εκ νέου στο μέλλον τα ζητήματα αυτά που άπτονται των οργανισμών αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δύο κύρια θέματα για τα ζητήματα που αναφέρθηκαν. Προς την κυρία Γκρέσλε, ζητώ συγγνώμη που δεν απάντησα σε σχέση με την ερώτηση όσον αφορά τη Γενική Γραμματεία. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο ενίσχυσης για φέτος. Πέρσι υπήρξε μια προσαρμογή στην αναδιοργάνωση με τη δημιουργία του Αντιπροέδρου και η Γενική Γραμματεία ενισχύθηκε μέσα σε αυτό το πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών προς τους νέους ε, αντιπροέδρους ε, που δεν έχουν ε, γενικούς, γενικές διευθύνσεις υπό αυτούς. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο, ας το πω έτσι, ξεχωριστό σχέδιο, γι' αυτό δεν απάντησε αυτό το ερώτημα. Όσον αφορά τους οργανισμούς και υπηρεσίες, μείωση 5% συνολικά, πώς να αντισταθμιστεί. Είχε συμφωνηθεί σε μια διοργανική συμφωνία αυτή η περικοπή. Αν θα συμφωνούσαν με διαφορετικό τρόπο για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα προσαρμόζαμε αυτή την προσέγγιση. Υπάρχει όμως μια διοργανική συμφωνία. Έχουμε και ένα διοργανικό σώμα και δεν ήταν δυνατόν να συνέλθει αυτό το όργανο μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια νέα ημερομηνία όμως για τον, μέχρι τον Ιούλιο. Κάθε φορά υπήρχε καθυστέρηση συνάντησης. Δεν είναι έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς μας, διότι συμφωνώ όταν συζητούμε για τις υπηρεσίες και οργανισμούς χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, αλλά και μια προσέγγιση ανάλογα με τις ανάγκες πιο εξειδικευμένα. Τούτων λεχθέντων, αυτό που προτείνουμε σήμερα είναι μια ad hoc προσέγγιση. Είναι μια ανώτατη προτεραιότητα για μας και πρέπει να ενισχυθούν αυτοί οι οργανισμοί. Προτείνουμε ένα δίκτυο ενίσχυσης που θα δίνει όχι ίσως επαρκή πλαίσια ενίσχυσης αλλά πρόσθετα κονδύλια και δυναμικό που θα μπορέσει μέσω του προϋπολογισμού να διασφαλιστεί. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω στοχεύουμε στην, στην κατεύθυνση αυτού που επιθυμεί το Κοινοβούλιο να συμβαίνει συχνότερα και προσβλέπω στη συζήτηση που θα έχουμε ο κύριος Γκάερ και εγώ μέσα στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού στις συζητήσεις μας. Merci. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Γκάρδια θα είστε η συγγήτρια για το ζήτημα αυτό. Μπορείτε να πάρετε το λόγο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Μέχρι τις 5 Ιουνίου το αργότερο θα πρέπει να κατευθούν τροπολογίες. Τα 5 15 Ιουνίου διορθώνει ο Πρόεδρος. Επομένως έχετε τρεις εβδομάδες περίπου στη διάθεσή σας. Alors nous revenons en arrière sur le point 8. Επιστρέφουμε στο σημείο 8. Κινητοποίηση του Ταμείου Ελληνικής Ευρωπαϊκή Ένωση, πλημμύρε στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Ιταλία. Ο κύριο Μορεζάνου, εισηγητής, και έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Συζητήσαμε σε σχέση με αυτό το θέμα πρωτού περάσουμε στο 5 ε, πράγματι συνδέεται αυτό με αυτή την έκθεση και εγώ όμω ε, θα πρέπει να παρουσιάσω αυτή την έκθεση σήμερα. Ουσιαστικά αυτή η έκθεση είναι η πρώτη κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης ε, όσον αφορά μέχρι το 2015 αφορά πλημμύρες στην Ιταλία, Βουλγαρία και Ρουμανία πέρσι. Το συνολικό ποσό που θα κινητοποιηθεί μέσω αυτής της απόφασης είναι 66,5 εκατομμύρια ευρώ. 56 θα στοχεύσουν στην Ιταλία, 8 εκατομμύρια Ρουμανία, 8,5 εκατομμύρια στη Ρουμανία και ε, τα υπόλοιπα δύο στην, ε, στην ε, τρίτη χώρα. Δημιούργησαν σημαντικές ζημιές αυτές οι πλημμύρες σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, γεωργία και υπήρχαν και θύματα. Έγιναν οι πλημμύρες ε, σε πέντε περιοχές στη Βόρεια Ιταλία. Οι συνολικές άμεσες ε, ζημιές ήταν 2, ε, κάτι δις, <clears throat> λιγότερα από τα 3, δις όσον αφορά την συνολική κατηγοριοποίηση για μίζωνα θεομηνία και έτσι βλέπουμε ότι καταχωρήθηκε ως περιφερειακή ε, ε, θεομηνία. Και σε σχέση με την Βουλγαρία χαρακτηρίστηκε ε, επιλέξιμη για τις περιφερειακές ζημιές που είχαν προκληθεί 79 εκατομμύρια ευρώ και το όριο για τον χαρακτηρισμό ως μείζων θεομηνία ήταν 232 γιατί η Ρουμανία υπήρχαν δύο αιτήματα. Ένα για τις αιαρινές ε, πλημμύρες ε, που ε, υπό τον όρο των ομόρων χωρών, δηλαδή με μίζωνες φυσικές καταστροφές στη γειτονική χώρα της Σερβίας για παράδειγμα. Και πάλι εδώ εντάχθηκε αυτό μέσα στο πλαίσιο των περιφερειακών θεομηνιών και 1,5% των άμεσων ζημιών θα μπορέσει να αποζημιωθεί. Προτείνεται η κινητοποίηση ενός συνολικού ποσού για αυτές τις ε, ζημιές και όπως ε, ανέφερε και η συγγήτρια προηγούμενα, ε, μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού έγκαιρα θα εγκριθεί ώστε οι τα κονδύλια αυτά να μπορέσουν έγκαιρα να έχουν αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Merci, Σας ευχαριστούμε κύριε Μουρεζάν. Από ό,τι φαίνεται δεν θέλει κανείς το λόγο. Κατάθεση τροπολογιών το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουνίου. Και στις 25 Ιουνίου θα γίνει η ψηφοφορία. Περνάμε στο σημείο 10, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Ο κύριος Ντεπχά έχει το λόγο. Έχει αναβληθεί, ο Πρόεδρος. Περνάμε στο σημείο 11 τότε. Ο κύριος Ντεβαντόφσκι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ και δεν έχουμε πολύ χρόνο και το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Έχει να κάνει με την μακροοικονομική ρεσιμότητα όσον αφορά την πολιτική συνοχή και τα διορθωτικά ταμεία. Πήγα σε διάφορες χώρες, κυρίως στις χώρες των καθαρών πληρωτών και πραγματικά τώρα πίστηκα ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η μακροοικονομική ρεσιμότητα και σε αυτά τα ταμεία. Στο παρελθόν χρησιμοποιούσαμε το κριτήριο αυτό μόνο για τα ταμεία συνοχή. Τώρα προτείνεται να καλυφθούν και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία επενδύσεων. Μα δίνει λοιπόν κατευθυντήριε γραμμέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου καλύπτεται μια συγκεκριματική δέσμη πολιτικών σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη δεν λάβουν την σωστή αντιμετώπιση όσον αφορά τη δικασία που Αυτό δεν καλύπτεται. Καλύπτεται η αδειοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ζητήσει τον επαναπρογραμματισμό κάποιων κονδυλίων, καθώς επίσης και την αναθεώρηση της Συμφωνίας Τερικής Σχέσης, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και στην οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση από τα κράτη-μέλη, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναστείλει και τι πληρωμέ προ τα κράτη-μέλη. Στην πρότασή μου λοιπόν, στην γνωμοδότησή μου προ την Επιτροπή Περιφερειακής ανάπτυξη, είναι να εγκριθεί ο κανονισμός αυτός, άλλωστε Μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε κάποιε αποφάσει, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν θα πρέπει να τιμωρούμε τελικά περιφερειακέ οργανώσει επειδή το κεντρικό κράτο δεν έχει συμμορφωθεί επαρκώ. Είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε, αλλά χρειαζόμαστε και ένα καλύτερο διάλογο με τα κράτη-μέλη, γιατί μιλάμε εδώ πέρα για επιμερισμένη τελικά ευθύνη. Πολύ συχνά αναφερόμαστε σε πολιετή εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία δεν συνάδουν με τον πολιτή χαρακτήρα που μπορεί να έχουν κάποια προγράμματα της πολιτικής συνοχής. Και στη συνέχεια έχουμε και τον ετήσιο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει τα όσα προβλέπονται στο κείμενο αυτό να αποτελούν ίστατη λύση η οποία θα χρησιμοποιείται αναλογικά και πολύ προσεκτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι τελικά μπορεί να υπονομεύσει την προβλεψιμότητα της πολιτικής συνοχής καθώς επίσης και τον προγραμματισμό όσον αφορά τα κονδύλια και θα πρέπει βέβαια να εμπλακεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2017 θέλουμε και μια έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Τα είπα εν συντομία, αλλά νομίζω ότι κάλυψε τα σημαντικότερα σημεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λεβαντόφσκι, σας ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις αυτές, για το ότι ευσύνοπτα παρουσιάσατε τα επιχειρήματά σας. Δεν θέλει κανείς το λόγο, δεν υπάρχει καμία παρατήρηση. Θα επανέλθουμε στο σημείο αυτό. Και περνάμε στο τελευταίο σημείο της της διάταξης. Ο κύριος Μικάλη Μπερζέκ προσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά μια έκθεση για την οποία είχαμε ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Μια έκθεση την οποία εξετάσαμε στην Επιτροπή μας στις 6 Μαΐου και είχε να κάνει με έναν νέο συνεργάτη, σύμβουλο που θα χρησιμοποιούσαν οι επίτροποι, ένα επίτροπο. Θα θέλαμε σχετικά με την πρόταση αυτή περισσότερε πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε την αλλαγή απόψεων. Ο κύριο Μπερζέ έχει το λόγο. Στη en effet rien ε, είχαμε θίξει αυτό το ζήτημα. Ο κύριο Δεπρέ, αν θυμάμαι, εκείνη την ημέρα είχε ζητήσει διευκρινήσει. Όχι, έτσι δεν είναι, κύριε Δεπρέ? Εγώ έτσι νομίζω ότι είχαμε πει τότε. Υπήρχε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ιδιαίτερη περίπτωση ενός συμβούλου για ειδικέ εκστρατείες, για δημόσιες σχέσεις που θα βοηθούσε έναν επίτροπο για την πρόθεση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα ή στις χώρες εκείνες που γνωρίζει καλύτερα ο Επίτροπος. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζουμε λίγα περισσότερα πράγματα όσον αφορά τη νέα αυτή θέση και το πώς αιτιολογεί τη δημιουργία της νέας αυτής θέσης, η νέα αυτή πρόσληψη. Πώς μπορεί να μας απαντήσει ο υπεύθυνο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, ποια είναι η νομική βάση για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Αναφέρομαι εδώ πέρα στο καταστατικό του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφερόμαστε στο άρθρο 123 παράγραφος 2 του καταστατικού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο για την πρόσληψη δικών συμβούλων πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση με την αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή προτού υπογραφεί η σύμβαση πρόσληψης του νέου του συμβούλου. Γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων με εσά ως αρχή αρμόδια για τον προπολογισμό. Η διάταξη αυτή υπάρχει από το 1962 και στόχος της διάταξης αυτής είναι να αντισταθμίσουμε πολλές φορές το ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους υπαλλήλου, το μόνο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το λοιπό προσωπικό και τους ειδικού συμβούλους από την άλλη. Ξέρετε ότι υπάρχει συγκεκριμένη κλίμακα μισθοδοσία όσον αφορά το λοιπό προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώ το μόνο προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη όμω δεν έχουμε συγκεκριμένη κλίμακα μισθοδοσία όσον αφορά του ειδικού συμβούλου που απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό ακριβώ το λόγο προβλέπεται στην κοινοτική νομοθεσία ότι η αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή έχει τη δυνατότητα να εξετάζει και να ελέγχει τη σκοπιμότητα πρόσληψης Ενό ειδικού συμβούλου και αν ο άνθρωπος αυτός λαμβάνει τη σωστή μισθοδοσία, τις, σωστές αποδοχές και αν δικαιολογούνται αυτές οι επιπλέον αποδοχές. Η ανταλλαγή λοιπόν αυτή απόψη έχει να κάνει μόνο με τις αποδοχές του ειδικού αυτού συμβούλου, δεν έχει να κάνει με τη γενικότερη πολιτική που διέπει το προσωπικό και το λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος Διακόπτη. Με άλλα λόγια αναφερόμαστε εδώ πέρα σε μια διαδικασία που δεν είναι ιδιαίτερα λογική, είναι μια καθαρή τυπικότητα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι. Επί της ουσίας δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Όχι, θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω για το τι προβλέπετε, Πρόεδρος. Όχι, μας έκανε εντύπωση ότι ο Επίτροπος ζητά την πρόσληψη ειδικού συμβούλου για να εξηγήσει τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα που ο Επίτροπος γνωρίζει καλύτερα για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή να γίνει διαβούλευση με την Επιτροπή Προπολογισμών. Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αναφερθώ σε δύο-τρία πράγματα με την αδειά σα. Όσον αφορά το άρθρο 123 παράγραφος 2 του καταστατικού του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους ιστορικούς κανόνες Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπονται τρία επίπεδα, α9, α12, πρόεδρος διακόπτη, όλα αυτά είναι καθαρά διοικητικά, γραφειοκρατικά, έχουμε τόσα άλλα σημαντικά πράγματα να καλύψουμε, πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να δαπανίσουμε χρόνο για το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστούμε πάντως για τα στοιχεία τα οποία μας δώσατε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή όμως να κάνουμε κάτι το ουσιαστικό. Κύριε Ντεπχέ και οι υπόλοιποι συντονιστές νομίζω ότι έχετε καλυφθεί, έτσι δεν είναι, από τα στοιχεία που ακούσατε. Δεν Νομίζω ότι καλούμεθα τώρα εμεί αυτή τη στιγμή με τέτοιε λεπτομέρειε να ενημερωθούμε για το πόσα χρήματα θα λαμβάνει ένα ειδικό σύμβουλο μια τέτοια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ανεφλόγου και ουσία. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι απαντήθηκαν οι οδήποτε ερωτήματα μπορεί να είχαν οι συντονιστέ. Ολοκληρώσουμε την μερίσια διάταξη. Άλλε ερωτήσει, όχι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αύριο το πρωί συνεδριάζουμε. Είναι πολύ σημαντική η συνεδριασή μας, καθότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα να με ενημερώσει για το σχέδιο προπολογισμού 2016. Κύριε Ντεπχά, θέλετε το λόγο. 10 η ώρα αύριο. Στις 10 η ώρα αύριο το πρωί. Σε αυτή την αίθουσα ρωτάει ο Πρόεδρος. Όχι, θα ήταν πολύ απλό να ήταν έτσι. Μάλιστα, καλό σας βράδυ.